Bueno. Bien, queridos colegas, vamos a comenzar la sesión de esta tarde. Καλώς συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να πω εδώ ότι ο κύριος Πρόκ είναι αδιάθετος μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα να πω ότι το briefing το οποίο θα έπρεπε να γίνει για την επίσκεψη στη ΣΥΠΑ δεν μπορεί να γίνει βέβαια. Ε, να πω επίσης ότι η αντεπροσωπεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν θα συζητηθεί σήμερα. Έχουμε ένα νέο σημείο, την έκθεση Κουκάνα για τη διακοινοβουλευτική ε, συνάντηση που έγινε στην Αλβανία. Η ενημέρωση της κυρίας Κοστέλο για την Παλαιστίνη έχει αναβληθεί και αυτή γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να είναι παρούσα. Πρόεδρε, σχετικά με την Παλαιστίνη, εγώ μόλις επέστρεψα από εκεί ε, με την αντιπροσωπεία. Αν θέλετε μπορώ να σας ενημερώσω. Προφορικά βέβαια μπορώ να σας δώσω μια περιγραφή του τι συνέβη εκεί. Γιατί είναι στην επικαιρότητα τα θέματα τα Παλαιστινιακά και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος γι' αυτό. Ευχαριστώ, θα λάβουμε υπόψη μας την διαθεσιμότητά σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν τα μέλη της Επιτροπής δεν ξέρω αν νομίζετε ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό κυρίως ε, με την παρουσία της Προέδρου της Αντιπροσωπείας. Αν όχι μπορούμε να το συζητήσουμε όπως είπε ο κ. Σάρκινς. Λοιπόν, πέρα από αυτά δέχεστε την ημερήσια διάταξη, εντάξει. Το πρώτο θέμα είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρας και της Τετάρτης Σεπτεμβρίου. Ξέρετε ποια είναι η διαδικασία. Και φτάνουμε στο σημείο υπαρίθμου 4, την έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κλάδο αυτό. Ο κύριος Κουκάν είναι ο εισηγητής μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους οι περισσότερες από αυτές είναι πολύ χρήσιμες και συμμετέχουν θα έλεγα στη βελτίωση της έκθεσης. 346 συνολικά τροπολογίες. Τις εξέτασα με ρεαλιστικό τρόπο. Είχα και μια χρήσιμη συζήτηση με τους σκιώδεις τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για την επικοδομητική του στάση. Έχουμε προετοιμάσει εδώ 27 συμβιβαστικές. Ε, θα ήθελα να υπάρξει στήριξη για όλες τις συμβιβαστικές, αν και κατανοώ βέβαια ότι θα είναι δύσκολο για κάποιες ομάδες να υποστηρίξουν κάποιες από τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Σχετικά με τις θέσεις των ομάδων γύρω από τις τροπολογίες και συμβιβαστικές τροπολογίες, όπως είχα πει και στην πρώτη παρουσίαση που είχα κάνει, δεν είχα πρόθεση εγώ να δημιουργήσω μια έκθεση που να έχει τα πάντα. Ήθελα απλά με αρεαλιστικό τρόπο να υπογραμμίσω τα πιο σημαντικά θέματα και τις εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκέντρωσα σε θέματα τα οποία πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, ήταν στον πυρήνα των συζητήσεών μας, όπως η διασύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, ή τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες μετάβασης και το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων. Η ιδέα αυτή υποστηρίχθηκε από τα μέλη κατά τη διάρκεια της Επιτροπής, της συνεδρίασης της αρμόδιας υποεπιτροπής και υποστηρίχθηκε σαν ιδέα και από τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Το πρώτο τμήμα είναι το πλαίσιο, το δεύτερο είναι οι διαδικασίες μετάβασης και το τρίτο είναι στήριξη στα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Συνοπτικά θα περάσω ανάμεσα ε, στα σημαντικά σημεία αυτών των τριών τμήματων. Καταρχάς ένα οριζόντιο θέμα θα έλεγα, ένα θέμα που περιλαμβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά του σεβασμού της ελευθερίας έκφρασης, ε, της ελεύθερης συνείδησης, και για την ελευθερία κίνησης επίσης αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά μέσω των τροπολογιών θα ληφθούν ακόμα καλύτερα υπόψη με τον σωστό τρόπο. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω τις επικαλύψεις. Ζητήθηκε επίσης να τεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών και μεμονωμένων περιπτώσεων στην πρόταση της έκθεσής μου. Εγώ προσπαθώ να περιοριστώ σε σχέση με τα παραδείγματα αυτά, να μην είμαι αναλυτικός. Όμως μετά από αρκετές συζητήσεις που είχα, συμπεριέλαβα αρκετές περιπτώσεις επιπλέον από αυτές που είχα συζητήσει πρώτα. Σχετικά τώρα με τις τροπολογίες, να πω πάντα ότι στο πρώτο πλαίσιο, παράγραφοι 10 με 24, οι περισσότερες τροπολογίες είχαν σαν στόχο θα έλεγα το να δώσουν λεπτομέρειες ε, για, στο κείμενο για τους εκπροσώπους μας στον τομέα αυτό και για τον ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εταιρικέ συμφωνίες. Ε, προτείνω λοιπόν αρκετές συμβιβαστικές τροπολογίες που δεν δημιουργούν πρόβλημα μια νέα παράγραφος από τις τροπολογίες 94, 95, 97 και 98. Ζητάμε επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιότητα και κοινοβουλευτικός έλεγχος στις στρατηγικές αναχώρα. Στον συγκεκριμένο αυτό τομέα υπάρχει και μια τροπολογία σχετικά με την παρούσα ε, ε, έρευνα των συμπεριφορών του NSA και ζητώντας ε, να σταματήσουν ε, οι, εμπορικές, ε, οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτή την τροπολογία δεν μπορώ να την στηρίξω. Σχετικά με την τροπολογία που αφορά το επιχειρήν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά μπορώ να θέσω τα θέματα αυτά στην έκθεσή μου αλλά θα ήθελα από αυτούς που προτείνουν τις τροπολογίες αυτές κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Για τις ε, διαδικασίες μετάβασης προτείνω 12 συμβιβαστικές. Αυτές που θα συζητηθούν κυρίως αφορούν συγκεκριμένες χώρες. Μέσω των συμβιβαστικών προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε καλύτερα τις παραγράφους που αφορούν τη Συρία και την ε, Αίγυπτο, την Κίνα και την Ρωσία και δημιουργήσαμε και δύο νέες παραγράφους για το Θιβέτ και την Κούβα. Στην περίπτωση της Ρωσίας και της Κούβα οι συμβιβαστικές τροπολογίες αναφέρουν σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις παραβίασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μακνίτσκι, Πολιτόσκαγια, Σβαλοπάγια. Σχετικά τώρα με τις υπόλοιπες τροπολογίες. Υπάρχουν πολλές οι οποίες προσθέτουν παραγράφους για συγκεκριμένες χώρες και για εδάφη που ανησυχούν όπως Σαχέλ, Κασμίρ, Δυτική Σαχάρα, Κολομβία και Χιλή. Εγώ θα ασχοληθώ με τις τροπολογίες αυτές κατά περίπτωση και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζητήσεις. Υπάρχει επίσης και το θέμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εδώ νομίζω ότι απαιτείται να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση για να δούμε αν πράγματι ένα τέτοιο θέμα θα συμπεριληφθεί. Υπάρχουν ε, ομόλογες θα έλεγα τροπολογίες 2.85 και 2.88 που ζητούν επίσης να υπάρξει μία επιπλέον παράγραφος για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τις υποστηρίζω. Για το τελευταίο τμήμα της έκθεσης, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εννέα τροπολογίες καλύπτουν διάφορα θέματα όπως το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Ποινικό, η θανατική ποινή, ε, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, οι διακρίσεις και οι ε, επιτροπές παρατήρησης των εκλογικών διαδικασιών. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες δεν περιλαμβάνουν προβλήματα και τις συμπεριλαμβάνουμε στο κείμενό μας. Ε, δημιουργούνται κάποιες συμβιβαστικές επιπλέον για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, για την λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και για τα δικαιώματα των παιδιών. Αναφέρομαι επίσης και σε θέματα της έκθεσης όπου προσπαθήσαμε να βρούμε νέες συμβιβαστικές λύσεις στις περαιτέρω συζητήσει μας, όπου αυτό δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι τώρα. Θα σας ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά. Άκουσα ότι ότι κάποια σκιώδηση συγγήτρια από μια πολιτική ομάδα της Άλντε, αν κατάλαβα καλά, δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα και θα στείλει τα σχόλια της γραπτός, θα τα λάβω υπόψη μου ως να είτο παρούσα. Τίποτα άλλο. Eh, Ευχαριστώ τον κύριο Κουκάν. Θα δώσω το λόγο τώρα σε αυτούς που το ζήτησαν. Η κυρία Κοπά πρώτη. First of all, I Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδιαίτερο στον κύριο Κούκαν για την σύντομη αλλά περιεκτική δήλωσή του. Η έκθεσή του δίνει ένα καθαρό μήνυμα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προτεραιότητες. Πλαίσιο της πολιτικής, υποστήριξη από την Ένωση και ε, για τις ε, άλλες χώρες. Βέβαια υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία δεν αναφέρονται. Τουλάχιστον αυτό επισημαίνει η πολιτική μου ομάδα. Ή δεν αναφέρονται καθόλου ή δεν αναφέρονται επαρκώ. Και εκεί στοχεύουν οι τροπολογίες μας. Ένα σημαντικό μέρος των τροπολογιών μας αναφέρεται σε αυτούς που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, κοινωνία των πολιτών καθώς και στην παγκοσμιότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων διότι υφίστανται επιθέσει τέτοια πρόσωπα καθώ και περιορισμού στην κοινωνία των πολιτών. Και αυτό συναντάται σε πολλές χώρες και ίσως μακροπρόθεσμα είναι το πλέον επικίνδυνο στοιχείο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα περισσότερο μάλιστα φέτος από ό,τι προηγούμενα χρόνια. Δυσφημίσεις και καταδίκες για δίθεν δυσφημίσεις κλπ. καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών που αποδείχθηκε επικοδομητική, οι περισσότερες από τις συμβαστικέ τροπολογίες του εισηγητού κρίθηκαν επαρκείς και όπου σημειώθηκαν κάποια θέματα γρήγορα ε, συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τους πράσινους να μην ξεχωρίσουμε το πολιετές πρόγραμμα πλαίσιο. Σε, σε μια συμβιβαστική τροπολογία είχαμε ένα πρόβλημα με την κοπτική χριστιανική ε, κοινότητα αντί να μιλήσουμε για την ανεξιθρησκεία που θα ήταν γενικότερο. Καταφέραμε ωστόσο να συμφωνήσουμε και η θέση μας έγινε δεχτή. Και αναμένουμε τώρα τη νέα συμβαστική τροπολογία. Στην 13 συμφωνήσαμε να αναφερθούμε στη Συρία όχι ως Συριακή κρίση αλλά με βαρύτερη ορολογία διότι ξεφεύγει πολύ από τα όρια της κρίσης η κατάσταση εκεί. Για διάφορε τροπολογίε τώρα που ε, είχαμε από τη δική μα πολιτική ομάδα για το ICC προτείνουμε δεύτερη παράγραφο στην τροπολογία 14 που θα περιλάβει ορισμένες, ε, ορισμένα τμήματα από άλλε τροπολογίε, όπω 252, 258, 259 και άλλε για την ατιμορρησία καθώ και για την ε, παγκοσμιότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γίνανε δεκτές οι προτάσεις μας και γι' αυτό αναμένουμε τώρα τις νέες τροπολογίες του εισηγητού. Στη συμβαστική 23 το ίδιο πρόβλημα με την ε, συγκεκριμένη αναφορά σε χριστιανικές κοινότητες, ενώ εμείς προτιμούμε να αναφέρεται η ανεξιθρησκεία, η ελευθερία άσκησης θρησκευτικής συνείδησης. Για την 25 θα θέλαμε να υπάρξουν περισσότερες παραπομπές στα δικαιώματα των παιδιών. Δεν μας αρκεί η απλή ε, αναφορά τέτοιων θεμάτων, η απλή απαρίθμηση τέτοιων θεμάτων. Αναμένουμε μια διαφορετική τροπολογία από τον εισηγητή και να αναφέρεται ιδίως ε, στα παιδιά στρατιώτες καθώς και σε παιδιά τα οποία ε, κατηγορούνται ως μάγοι ή μάγισσες. Επίσης άλλα σημαντικά θέματα που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε εκτός για τις τροπολογίες που δεν περιλήφθηκαν στις συμβαστικές και θα ψηφιστούν ξεχωριστά υπάρχουν ορισμένα θέματα για μας ένα από αυτά είναι τα, τα μη επιδρομένα αεροσκάφη που είπε και ο κύριος Κούκαν. Η σωστή χρήση των οποίων είναι για την πολιτική ομάδα πολύ ε, σημαντική και βεβαίως η στρατιωτική τους χρήση σε χώρες όπως το Πακιστάν. Και δεύτερο, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η ομάδα μου στα δικαιώματα γυναικών και παιδιών διότι η έκθεση δεν αποδίδει τη σημασία που θα θέλαμε στα θέματα αυτά. Άρα δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένες, αλλά επιμένουμε να ψηφιστούν ορισμένε τροπολογίες μας ξεχωριστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τονίσουμε τη σημασία των θεμάτων που, στα οποία αναφέρονται. Πάντως ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Κούκαν για τη διάθεση συνεργασίας και το ανοιχτό του πνεύμα στη συζήτηση για τις σημαντικές τροπολογίες και σας ευχαριστώ και πάλι. Eh, Ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκανα για αυτή την, ε, αυτό το καλό προσχέδιο έκθεσης. Ε, είναι καλά εστιασμένη ε, και αφορά ακριβώς προτεραιότητες και όχι μια σειρά ασχέτων πραγμάτων εν είδη shopping list. Είχαμε επικοδομητικό διάλογο και καλές συμβαστικές λύσεις και από την πλευρά της δικιάς μου ομάδας ε, μπορώ να πω ότι στηρίζουμε αυτές τις ε, συμβαστικές λύσεις πλην του συμβιβασμού 2 η κυρία Κοπά αναφέρθηκε ήδη στο θέμα αυτό. Ε, πρόκειται για την ε, χρηματοδοτική οικονομική στήριξη ε, του Ευρωπαϊκού Εργαλείου για την Δημοκρατία και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εξ αρχής, ε, όταν είχαμε καθορίσει το πλαίσιο, είπαμε ότι δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να ε, βγουν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τη Δημοκρατία ε, και να μπουν σε κάποιο άλλο στοιχείο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Όταν γίνεται λόγος για στήριξη, ενωσιακή στήριξη, αυτό συμπεριλαμβάνει και τα κράτη επιμέλεια αφορά το 8, ε, αφορά το σχέδιο GSP Plus ε, και θα θέλαμε να γίνει η εφαρμογή ανά χώρα και νομίζω ότι με αυτή την προσέγγιση συμφωνούν ή μάλλον θα ψηφίσουν σήμερα οι συνάδελφοι της ΙΝΤΑ. Ε, γιατί ε, εάν θέλει κανείς ε, να ελέγξει πραγματικά το ε, GSP Plus και δεν έχει αναφορά αναμεμονωμένη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει την κατάσταση όσον ή το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ήταν για το συμβιβασμό υπαριθμών 8. Λίγο πιο μετά, στην ίδια παράγραφο, θα θέλαμε να πούμε το εξή. Ε, λέμε ε, να ελέγχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις, ε, διαδικασίε διαδικασίες επιτήρησης και αυτό να γίνεται μέσω ευραίων διαβολεύσεων με την τοπική κοινωνία των πολιτών, το Κοινοβούλιο της χώρας, καθώς επίσης και όλους τους πρωταγωνιστές σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είχε βγει από το κείμενο, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξαναμπεί. Εν τέλει, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κούκαν για τη στήριξη των τροπολογιών που αφορούν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καθώς επίσης ε, και την ε, ε, αναφορά σε μη επανδρομένα αεροσκάφη και επίσης όσον αφορά το κεφάλαιο της επιχειρηματικότητας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα να πω ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και στη συνέχιση προς αυτή την κατεύθυνση και ευχαριστώ τον κύριο Κούκαν για το πολύ καλό προσχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λεκμπίρελ. Κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι η παρούσα έκθεση δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη για τον συντάκτη της και γι' αυτό με πάρα πολύ μεγάλη χαρά βλέπω ότι ο κύριος Κουκάν πράγματι έχει πετύχει πάρα πολλά στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκθεσης του. Θα ήθελα να κάνω ένα, κάποιο, ένα πρώτο σχόλιο και για αυτά τα οποία είπε η προηγούμενη ομιλήτρια η κυρία Κοπά σχετικά με τους κόπτες της Αιγύπτου. Έχω την αίσθηση ότι η συγκεκριμένη αναφορά στην κοπτική μειονότητα δεν είναι αντίθετη με τις γενικότερες πρωτοβουλίες στις οποίες παραπέμπει ο εισηγητής στον τομέα των θρησκευτικών ελευθεριών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπογραμμίσει το συγκεκριμένο κλάδο, το συγκεκριμένο τομέα καλύτερα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κοκάν για την καλή του έκθεση, μια έκθεση ισορροπημένη πάνω σε ένα θέμα το οποίο όπως ε, ε, λέμε ε, κατέχει ένα κεντρικό σημείο εν πάση περιπτώσει στην ευρωπαϊκή προβληματική της εξωτερικής μας πολιτικής τίθενται θέματα θεμελιώδη, θεσμικά θέματα και ιδιαίτερα για τις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης και πρέπει να τροφοδοτήσουν ε, τις σκέψεις μας στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποια θέματα λοιπόν τα οποία πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής μας γενικότερα. Δεν ξέρω ακριβώς τις συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες έχει προετοιμάσει ο κύριος Κουκάν, αλλά θα τις μελετήσουμε με πολύ προσοχή και συγχαίρω εκ νέου τον κύριο Κουκάν για την τεράστια προσπάθειά του. Ευχαριστώ κύριε Μιγιάν. Ο κύριος Κουκάν παρακαλώ να κλείσει με τα τελικά του σχόλια την συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που μετήχαν στη συζήτηση. Αυτή βεβαίως δεν ήταν εύκολη έκθεση και είναι δύσκολο να διατυπωθεί με τρόπον ώστε να γίνει ε, ευνοϊκά αποδεκτή από όλους, αλλά στόχος μου είναι να βρω την ευρύτερη δυνατή ε, στήριξη, ε, γιατί με τον τρόπο αυτό βεβαίως το βάρος του εγγράφου είναι και πιο σημαντικό και μπορεί να επηρεάσει και την εικόνα που έχουμε προς τα έξω. Η, η παράγραφος που ανέφερε η κυρία Κοπά και η κυρία Λοχμπίλερ. Όπως είπα, και στην αρχική μου εισήγηση είμαι απολύτως διατεθειμένος να συνεχίσω τη συζήτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, φτάσουμε, να επιτύχουμε μία διατύπωση την οποία να μπορούμε και οι δύο πλευρές να αποδεχθούμε. Όσον αφορά τώρα ε, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, όσον αφορά και το ε, συμβιβασμό 10 που αναφέρθηκε προηγουμένως, βεβαίως μπορούμε να ξαναδούμε τα σημεία αυτά. Ε, ε, θα είμαι διαθέσιμος και ε, προς τους σκιώδεις και ανοιχτός σε προτάσεις έτσι ώστε η Επιτροπή μας να επιτύχει το μέγιστο δυνατό βαθμό ενότητας επί της εκθέσεως αυτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Με την παρέμβαση αυτή λοιπόν κλείνουμε την συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, για την έκθεση του κυρίου Κουκάν. Θα προχωρήσουμε στην εξέταση λοιπόν στο Στρασβούργο, ε, ή μάλλον τα, τις συμβιβαστικές τροπολογίες είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό γιατί τίθεται το θέμα υποσυζήτηση και στο Συμβούλιο Υπουργών σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και πόσο επηρεάζεται και επηρεάζει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα επιτρέψει να γίνει όχι μόνο μια αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2012, αλλά ε, γιατί ε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα και με τον κύριο Λαμπρινίδη, τον υπεύθυνο στην εξωτερική πολιτική για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, η προθεσμία είναι 21 Νοεμβρίου και έτσι θα μπορέσουν τα μέλη να ξεκαθαριστούν οι θέσεις και να κατατεθούν οι τροπολογίες. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλες συζητήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Θα περάσουμε στο 5 το debriefing για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 68η συνεδρίαση της Ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρχαν εκεί ο κύριος Λάκβιτ, Μιγιάν, Μάρτιν, Σούλτς, Μαρτίνι. Είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, να συναντηθούν με στελέχη των Ηνωμένων Εθνών και με τον ίδιο Μπαν Κιμούντ, τον δεύτερο γραμματέα, τον κύριο Φέλντερ, τον εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υπεύθυνη κυρία Κίνγκ για τον αφοπλισμό, ε, με εκπροσώπους της UNDP, της UNICEF, της ομάδας καταπολέμησης ε, της ε, τρομοκρατίας κτλ. κτλ. Συναντήθηκαν επίσης και με πολλούς εκπροσώπους κρατών μελών που συμμετέχουν στον Διεθνή Αυτό Οργανισμό, με τον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπους της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Παλαιστίνης. Προφανές είναι ότι η επίσκεψη της αντιπροσωπείας αυτή της Επιτροπής μας είχε να αντιμετωπίσει λόγω επικαιρότητα τα θέματα τα οποία τέθηκαν ιδιαίτερα στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή τη Συρία, τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως επίσης και τις κατασκοπικές δραστηριότητες οι οποίες ε, ε, υπογραμμίστηκαν στα πλαίσια της δράσης της NSA στις Ηνωμένε Πολιτείες. Η επίσκεψη αυτή είναι στην ουσία η συνέχεια μιας αντιπροσωπείας την οποία εμείς είχαμε στείλει στη Ουάσιγκτον τις προηγούμενες μέρες και που ασχολήθηκε με τα συγκεκριμένα θέματα. Για τη Συρία ε, θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο βασικά θέματα. Το ένα αφορά την διάλυση του χημικού οπλοστασίου οι υπεύθυνοι των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκαν στην, στο ύψιστο επίπεδο δυσκολίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσουν, να ανοιχνεύσουν, να εντοπίσουν και να καταστρέψουν τις συγκεκριμένες ποσότητες των χημικών όπλων και να μεταφερθούν μάλιστα και κάποια από αυτά τα χημικά όπλα εφόσον δεν μπορούν να, γίνουν, να γίνει η καταστροφή τους τοπικά και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και φυσικά οι πολιτικές διαδικασίες ειρήνευσης, οι λεγόμενες διαπραγματεύσεις της Γενέβης, οι οποίες όλοι γνωρίζουν ότι συναντούν τεράστιες δυσκολίες λόγω των πάρα πολύ μεγάλων διαφορών οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στις ε, διάφορες πλευρές, στις διάφορες συνιστώσεις καλύτερα της αντιπολίτευσης. Οι εκλεκτοί συνομιλητές μας με τους οποίους συναντηθήκαμε μας είπαν ότι το πρόβλημα μέσω της πολιτικής διαδικασίας δεν είναι κάτι το οποίο θα προκληθεί μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και οι λύσεις θα πρέπει να βρεθούν μέσω διμερούς διαλόγου ανάμεσα κυρίως στα Ηνωμένες, στις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσία. Εξέφρασαν ορισμένα κράτη-μέλη την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στην κατάσταση ε, η απόφαση που ελήφθη σε σχέση με τα χημικά όπλα δυστυχώς δεν επιλύει την ουσία, το πρόβλημα στην ουσία του, το συριακό πρόβλημα. Συνεχίζεται η βία με τρομερό τρόπο και αυτό περιπλέκει ακόμα περισσότερο, με φρικτό θα έλεγα τρόπο, την ανθρωπιστική κατάσταση η οποία δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες και παρεμποδίζει και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να μου επιτρέψετε να σας υπογραμμίσω τη σημασία που έχει το ότι όλοι οι συνομιλητές μας αναφέρθηκαν στην ανθρωπιστική παρέμβαση η οποία υποστηρίζεται και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσπάθειες τις οποίες κάνει ιδιαίτερα η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα. Νομίζω λοιπόν ότι ο βασικός κίνδυνος ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση έρχεται στην επιφάνεια είναι να μην συντονιστούν οι προσπάθειες που θα οδηγήσουν σε μια πολιτική λύση ε, ακριβώς λόγω των μεγάλων διαφορών που ε, υπάρχουν ανάμεσα στις ομάδες και στην μεγάλη δύναμη που έχουν οι Ισλαμιστές. Αυτό το υπογράμμισε και ο Ρώσος πρέσβης και πολλοί άλλοι συνομιλητές μας. Ε, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, τρομερές καταστάσεις για χώρες όπως η Ορδανία, ο Λίβανος και δεν θα πρέπει οι χώρες αυτές να γίνουν παράπλευρες απώλειες, να θεωρηθούν παράπλευρες απώλειες της κατάστασης στη Συρία. Θυμίζω ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιών επίσης θίγονται με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο από την συγκεκριμένη σύγκρουση Υπάρχουν επιδημίες ε, που φαίνεται να αναφαίνονται ιδιαίτερα στον τομέα της πολιομελίτιδας κτλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η προστασία των ιδιωτικών ε, στοιχείων και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και ψηφιακών ταυτοτήτων. Αυτό έγινε στα πλαίσια της αντιπροσωπείας μας ε, συζήτηση από αυτό, ιδιαίτερα στην Washington, αλλά και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ε, προτάθηκε να υπάρξει ένα ψήφισμα γύρω από το τομέα αυτό μετά από πρωτοβουλία της Βαζιλίας και της Αργεντινής. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο κατατέθηκε, προτάθηκε πρώτα από την Γερμανία και ζητήθηκε από τους πρέσβεις της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα μας είπαν ότι ε, επιφυλάσσονται να απαντήσουν ε, σε επίπεδο λεπτομεριών και θα είναι πάρα πολύ προσεκτική γύρω από το συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης σε καμία περίπτωση να μην λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένες δραστηριότητες σε σχέση με το διαδίκτυο. Το θέμα αυτό το αντιμετωπίσαμε και στα πλαίσια της συνάντησης την οποία είχαμε με την κυρία Ρέντινγκ που ήταν εκεί παρούσα και οι δικές της εντυπώσεις από την επίσκεψη κυρίως στη Washington ήταν ότι σε ένα πρώτο επίπεδο φαίνεται ότι υπήρξε μια χειροτέρευση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιοι, αυτό ήταν ξεκάθαρο σε κάποιες από τις συζητήσεις τις οποίες είχαμε και σε κάποια από τα μέλη της δικής μας επιτροπής που ήταν παρόντα και στη Ουάσιγκτον. Η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε μια επανεξισορρόπηση της παρακολούθησης των ιδιωτικών στοιχείων και ταυτοτήτων. Σχετικά τώρα για το άλλο θέμα, το της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έχουν υπάρξει σημαντικά βήματα προόδου εδώ. Υπάρχει μια στασιμότητα και ορισμένοι πιστεύουν ότι στα πλαίσια των 70 χρόνων της λειτουργίας του οργανισμού ίσως ο Γενικός Γραμματέας να ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία η οποία θα έχει σαν στόχο να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που έχουμε ε, αντιμετωπίσει σήμερα. Ε, υπάρχει μια γαλλική πρωτοβουλία η οποία έχει σαν στόχο να μην χρησιμοποιούν το δικαίωμα βέτο σε περιπτώσεις όπως η γενοκτονία στα πλαίσια των συνεδριάσεων και της λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι έντονες και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα σύντομα. Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι τα νέα μόνιμα μέλη θα πρέπει να έχουν μια περιφερειακή, να υπακούν σε μια περιφερειακή κατανομή. Άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε για να κλείσω αυτή τη σύντομη, πολύ σύντομη παρουσίαση ήταν το θέμα των διαφορών που υπάρχουν ε, σε επίπεδο Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με την κλίση του Προέδρου Κενιάτα ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θέλει να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει μια μορφή απόδοσης δικαιοσύνης σε διεθνές επίπεδο με δύο ταχύτητες, Ενθυμίστε ότι τον Νοέμβριο έγινε μια ψηφοφορία στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, τώρα αναφέρομαι στα της Παλαιστίνης, όπου πήρε ε, την, ε, τον τίτλο του μέλους πλέον η Παλαιστίνη. Συναντηθήκαμε με τον πρέσβη λοιπόν της Παλαιστίνης και με χώρες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Συζητήσαμε τα θέματα της ειρηνευτικής διαδικασίας και εδώ δυστυχώς δεν υπήρξαν πάρα πολλά στοιχεία αισιοδοξία. Είχαμε και ε, συναντήσεις όπως είπαμε τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών της ΥΠΑ της Αυμοστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τους εκπροσώπους της UNICEF, με τους εκπροσώπους της Επιτροπής για τις Γυναίκες, με τους εκπροσώπους της Ομάδας Δράσης ε, κατά της, ε, ε, κατά της τρομοκρατίας, όπως επίσης και της ε, σεξουαλικής βίας. Συζητήσαμε τα θέματα αυτά επί τη βάση του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός εισφορέας αν θέλετε στις προσπάθειες οικονομικά όλων αυτών των οργανισμών. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό εδώ να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπό μας στα Ηνωμένα Έθνη και στους συνεργάτες του, ε, τον κύριο Μαξ Άντερσον Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής μας θα πρέπει να στείλει μία επιστολή για να ευχαριστήσουμε την υπηρεσία μας εκεί και για τις συνθήκες οι οποίες ε, διαμορφώθηκαν πολύ ευνοϊκές. Ο κύριος Μιγιάν Μοντ θέλει το λόγο για να κάνει και αυτός τις δικές του παρατηρήσεις και σχόλια. Έχει το λόγο ο κύριος Μιγιάν Μοντ. Ευχαριστώ και εγώ σαν μέλος της αντιπροσωπείας Presidenta, lo que usted ya nos ha contado de esta delegación que usted mismo finalmente tuvo que presidir. Eh, yo quizá destacaría sobre todo... Porque... Eh, λοιπόν, ε, σε τέτοιου είδους ταξίδια έχω θα έλεγα πάρα πολύ μεγάλη πείρα, έχω πάει επανειλημμένα και νομίζω ότι οι συναντήσεις που έγιναν αυτή τη φορά ήταν στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Ε, μας, μας υποδέχθηκε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο στο παρελθόν. Και δεν υπήρξε μια συνάντηση απλά σε επίπεδο πρωτοκόλου, είχαμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις, ε, μας έκανε δεκτούς επίσης και ο δεύτερος Γενικός Γραμματέας και τέλος, εν πάση περιπτώσει, συναντήσαμε ένα μεγάλο αριθμό μελών των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι όλοι διαμορφώσαμε μια αντίληψη σε σχέση με τη λειτουργία των Ηνωμένων Εθνών και είδαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να υπάρξει η δυνατότητα ε, καλύτερης εταιρική σχέσης ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Νομίζω ότι ο πρόεδρος μας, ο κύριος Σαλαφράνκα, είπε και για τη συνάντηση με τον Ρώσο πρέσβη. Είναι η πρώτη φορά που γίναμε δεκτοί. Είπαμε επίσης ότι είχαμε προηγούμενες συναντήσεις και με τον Γάλλο πρέσβη. Νομίζω ότι θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι μας συνόδευαν και την γραμματεία γενικότερα. Να συγχαρούμε επίσης και τον πρέσβη μας εκεί, ο οποίος μας βοήθησε ιδιαίτερα όπως ακριβώς και τα είπε ε, ο κύριος Σαλαφράνκα ε, και η συνάντηση με την κυρία Ρέντινγκ επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρουσα η συνάντηση αυτή και για το επίπεδο στο οποίο έγινε και για το ενδιαφέρον το οποίο παρουσίασε. Κύριος Δεμέρσμακερ είναι εδώ. Eh, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ήδη μας δώσατε μια εικόνα της επίσκεψης και συμφωνώ με τα όσα εξήγησαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές στη διάρκεια των ε, συναντήσεών μας κυρίως συζητήθηκε το δράμα της Συρίας και δυστυχώς αυτά που έμειναν στη μνήμη μου ήταν η απεσιόδοξη εικόνα που έδωσε, που μας περιέγραψε και η αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη και ο πρέσβης της Γαλλίας. Και τα δύο αυτά πρόσωπα είπαν ότι ουδής έχει τη λύση αυτή τη στιγμή. Ήδη η πολιτική λύση φαίνεται να είναι πολύ μακριά. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια, πρέπει να έχει υπόψη κανείς και το ενδεχόμενο κάποιων στρατηγικών επιπτώσεων και βέβαια αυτό που θυμούμαστε περισσότερο είναι οι εικόνες της Άντζελα Κέιν που μας ε, εξήγησε δηλαδή της ε, τρομερά σκληρής και δύσκολης δουλειάς που κάνουν οι διάφοροι οργανισμοί και άλλοι φορείς επιτόπου και σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό των χημικών όπλων, την μεταφορά των χημικών αυτών όπλων, την καταστροφή τους πρέπει να επισκεφθούμε δύο μέρη στην Συρία. Ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε τις πρόοδους που έχουν σημειωθεί σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και καταστροφή του χημικού προστασίου στη Συρία, αλλά πάντως γενικά η κατάσταση περιγράφεται με πολύ μελανά χρώματα. Για τη χρήση τώρα των μη επανδρομένων αεροσκαφών, γιατί μιλήσαμε και προηγουμένως για το θέμα αυτό και θα επισημάνω τα, είσαι, είπε, όσα είπε ο Ιμάν Σιμόνοβιτς που είναι εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο οποίος αναρωτήθηκε αν δεν θα πρέπει να ψηφιστούν διεθνείς κανόνες που να ρυθμίζουν τα της χρήσης των μη επανδομένων αεροσκαφών και σε καταστάσεις άλλες εκτός πολεμικών διότι αυτά τα αεροσκάφη γίνονται όλο και λιγότερο δαπανηρή χρήση τους δηλαδή και θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Αλλά αυτά απορρίφθηκαν από τον εκπρόσωπο των Ενωμένων Πολιτειών. Επίσης, κατ' επανάληψη τέθηκε το θέμα της λαοκρατικής δημοκρατίας του Κόγκο. Είμαι Βέλγος και με απασχολεί πολύ το θέμα της χώρας αυτής. Η κατάσταση στο Κονγκό και η βία, ιδίως σε βάρος των γυναικών, έχει γίνει πλέον έχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσεις. Πρέπει κάτι να γίνει επί τόπου και ίσως η νέα στρατιωτική κατάσταση εκεί προσφέρει κάποιες δυνατότητες παρέμβασης. Πάντως επανέρχομαι στα όσα είπε ο Πρόεδρός μας και δηλώνω και εγώ την ικανοποίησή μου για τις συζητήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των Ενωμένων Εθνών που μας είπε ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και υπέρ της αηφόρου ανάπτυξης που είναι και οι πρώτες προτεραιότητες των Ενωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχα σε τέτοια αντιπροσωπεία και για μένα πρόκειται για μια εμπειρία εξαιρετικά σημαντική και συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Σόλτ, Σόλτς, συγγνώμη, κύριο Σόλτς. Δεν έχει μικρόφωνο κύριο Σόλτ; Δεν ξέρω αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόλαβα να ακούσω όλη τη συζήτηση. Ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής για το πλούσιο πρόγραμμα των συναντήσεων που μας επέτρεψε να διεξαγάγουμε πραγματικά καρποφόρες συναντήσεις με πλείονες συνομιλητές από πλευρά των ΕΕ. και σημειώνω ιδιαίτερα ειδικά για τον ειδικό εισηγητή των ΕΕ Εθνών για την γενετήσια βία σε περιπτώσεις συγκρούσεων, που ήταν πολύ περίπλοκη και δύσκολη συνάντηση, γιατί ακούσαμε το τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και τονίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλει στη μείωση της βίας αυτής δεν πρέπει μόνο να συζητήσουμε αυτή τη γενετήσια βία στις συγκρούσεις, αλλά και μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ισότητας των φίλων και της δημοκρατίας. Διότι υπάρχουν και στοιχεία πολιτιστικών συγκρούσεων σε πολλές χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τονίστηκε από πλευρά, πλευρά των εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο Πεκίνο συνήκωση για θέματα γενετήσιας βίας και να δώσει μια νέα όθηση στη συζήτηση αυτή. Μου φάνηκε ενδιαφέρον ότι πλήρωνε από τους συνομιλητές μας μας τόνισαν και το ρόλο του ICC που θεωρούν ότι πρέπει να παίξει τον ρόλο του το, ποινικό, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και Ελπίζω δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της θα εκπληρώσουν, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα εκπληρώσουν τις υποχρώσεις τους και προβλέποντας και στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης mm. ώστε να έχουμε και ξεκάθαρες κατευθύνσεις για την εργασία μας για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Θα μείνω σε αυτά. Συζητήθηκαν και θέματα πυρηνικού αφοπλισμού καθώς και τις διαδικασίες καταστροφής των χημικών όπλων. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας κύριε Σόλτς. Κλείνουμε την υπόθεση αυτή. Να διευκρινίσω εδώ σχετικά με την έκθεση του κυρίου Κουκάν ότι 21η Νοεμβρίου δεν είναι η ημερομηνία κατάθεσης των απολογιών. Είναι η ψηφορία προβλέπεται για τις 14 του μηνός και ακριβώς επειδή καταργήθηκε η προηγούμενη συνεδρίαση θα, θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρία στην οποία ανάφερα. Εδώ να καλωσορίσω εκπροσώπους από τη Σομαλία και την Ουγκάντα που εκπροσωπούν τις Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Κοινοβουλίων τους. Τους εύχομαι μια κακοφόρο συνάντηση εδώ στις Βρυξέλλες su Ελπίζω να υπάρξει καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στι δικέ του και τι δικές μας εργασίε. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το debriefing από πλευρά του κυρίου Κούκαν για την έκτη συνάντηση σταθεροποίηση με την Αλβανία που γίνεται σε μια, ε, θα έλεγα, επίκαιρη στιγμή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά μας μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Πρόοδου και καλείται πλέον το Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση για την υποψηφιότητα της Αλβανίας ως υποψηφίας προς ένταξη χώρας. Η έκθεση λοιπόν την οποία θα μας παρουσιάσει ο κύριος Κουκάν θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, η κοινοβουλευτική συνεδρίαση έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες στα Τύρανα. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από 7 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Νικόλα Βουλιάνιτς ε, του ΕΛΚ, εισηγητής. Εφτά εβδομάδες λοιπόν έγινε πριν από το ε, Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στο οποίο θα αποφασιστεί εάν θα δοθεί το καθεστώς υποψηφιότητας ε, στην Αλβανία όπως προτείνει, συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κοινή κοινοβουλευτική λοιπόν συνεδρίαση έλαβε χώρα και ε, στην ολοκλήρωσή της ε, υπέγραψε κοινή συμφωνία σε κείμενο. Παρατηρούμε βελτίωση του πολιτικού διαλόγου. Πιο ειρηνικές ε, συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Το πολιτικό περιβάλλον, η πολιτική ατμόσφαιρα στην Αλβανία βεβαίως πόρο απέχει ε, το να είναι ικανοποιητική, όμως διαρκώς βελτιούται. Το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι βελτιώνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι εταίροι μας εκπροσωπούν όλο το πολιτικό φάσμα και ε, προχωρούν σε τελείως διαφορετική ανάγνωση των επιτευγμάτων των πρώτων 40 ημερών της νέας κυβέρνησης. Το σημαντικό ήταν ότι όλες οι πλευρές παρουσίασαν πολύ πιστικά επιχειρήματα ε, εκφραζόμενοι θετικά, υπέρ δηλαδή της, ε, του καθεστώτος ε, υποψηφιότητας πριν από τις τελευταίες εκλογές είχε γίνει αποδεκτό ένα κείμενο ε, σε συνενετική βάση. Διαφορετικές ερμηνείες αφορούν την θέση ισχύ ε, και την ε, απαραίτητη εφαρμογή νόμων ε, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τη νέα κατάσταση, δηλαδή η νέα αντιπολίτευση ε, κατηγορεί την νέα ε, κυβέρνηση για μαζικές απολύσεις και στη δημοσιοδιοίκηση και στην αστυνομία. Τη θέση των απολυμένων δε κατηγορούν, καταγγέλουν ότι παίρνουν προσκύμινη στην κυβέρνηση. Επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης βεβαίως γίνεται λόγος για απόλυση διεφθαρμένων και μη αποτελεσματικών υπαλλήλων. Ε, το θέμα είναι ότι η μαζική προσπάθεια μεταρρύθμιση έτσι όπως παρουσιάζεται από την νυν κυβέρνηση είναι βεβαίως απαραίτητη. Αλλά οι αλλαγές στο οργανόγραμμα των δημοσίων υπηρεσιών είναι υπερβολικά ε, μεγάλες έτσι ώστε να παραμένουν σε ένα, νομικό, ε, σε ένα νόμιμο πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε ε, απαλυφή της διαφθοράς, βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Ε, πρέπει να πούμε όμως ότι έγιναν πολλές επιδρομές αστυνομικές έτσι ώστε ε, να κλείσουν ε, παράνομα ε, να κλείσουν παράνομες λέσχες χαρτοπεξίας κλπ. Η Αλβανία έχει στη διάθεσή της ακόμα έξι εβδομάδες έτσι ώστε να πείσει ότι οι αλλαγές, οι, τροποποιη... μεταρρυθμίσεις της και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει οδηγούν ε, σε μια ε, επικοδομητική μεταρρύθμιση και όχι ότι πρόκειται για αλλαγές ε, οι οποίες γίνονται στο πόδι και οι οποίες αφορούν μονάχα το βόλεμα ημετέρων κτλ. Ε, βεβαίως θα πρέπει να ε, σημειώσουμε τις θετικές αλλαγές, οι οποίες όμως θα πρέπει να ακολουθηθούν από ουσιώδεις ε, ακόμα πιο θετικές αλλαγές. Φυσικά και ο χρόνος της νέας κυβέρνησης ήταν πάρα πολύ λίγος. Η κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει με συγκεκριμένες πράξεις ότι η ερμηνεία που δίνει για τα τεκτενόμενα είναι όντως θετική επισκεφθήκαμε την Αλβανία και μετά επισκεφθήκαμε και το Κωσυφοπέδιο. αλλά ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να τα μπερδέψουμε όλα. Το debriefing, η ενημέρωση για το Κωσυφοπέδιο πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Ε, υπήρξε επίσης και αποστολή παρατήρησης των εκλογών στο Κωσυφοπέδιο. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο ενημέρωσης. Ε, ευχαριστούμε κύριε Κούκαν, κύριος Μπουλιανίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Κόκαν έκανε μια σωστή περιγραφή του τι είδαμε εκεί. Πήγα εκεί σαν συνεισηγητής της Επιτροπής μας. Υπάρχουν βελτιώσεις προφανής στην κατάσταση στην Αλβανία. Υπήρξε όμως έλλειψη διαλόγου όχι μόνο ανάμεσα σε κόμματα, αλλά και ανάμεσα σε άλλους εμπλεκομένους θα έλεγα στην κατάσταση στη χώρα. Είχα πάει πριν δύο εβδομάδες, συναντήθηκα με συνδικαλιστές και εργοδότες, με τον Όμπουτσμαν και με μέλη του Κοινοβουλίου και διαπίστωσα ότι υπάρχει πάντα η προσπάθεια του να μεταφέρει κανείς την ευθύνη στην απέναντι πλευρά. Αυτή είναι μια γενική αντίληψη. Οπότε αυτό κάνει δύσκολο το πολιτικό διάλογο και γι' αυτό ο διάλογος χρειάζεται στην Αλβανία και εδώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βοηθήσει να το πετύχουν. Πολλά ακούστηκαν για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για το οργανωμένο έγκλημα κτλ ότι υπάρχει διαφθορά και έγκλημα το ξέρουμε αυτό και από τα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν και αρκετές στατιστικές που το αποδεικνύουν αυτό. Προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, να πάρουν κάποια μέτρα, έχουν ήδη πάρει κάποια μέτρα. Αν δει κανείς την κατάσταση στη χώρα ε, σχετικά με το πόσο έχουν βελτιωθεί θα διαπιστώσει κανείς ότι πράγματι η βελτίωση είναι σημαντική αλλά αν από την άλλη συγκρίνουμε την κατάσταση στην Αλβανία με την Ολλανδία ή με την Δανία, τότε είναι προφανές ότι δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Δεν είμαι βέβαιος αν πράγματι η πολιτική ελίτ της χώρας κατανοεί το τι ε, τους περιμένει. Εάν δεν τους βοηθήσουμε τώρα, γρήγορα εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσουν να συλλάβουν, θα έλεγα, την κατάσταση ε, σε ένα έφετο χρονικό διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Αλβανία είναι σοβαρή υποψηφία έτσι ώστε να θεωρηθεί το Δεκέμβριο υποψήφια προς ένταξη, ανεξαρτήτως του τι θα πει το Συμβούλιο. Ότι θέλει θα πει το Συμβούλιο βέβαια, αλλά πάντως η χώρα έχει παρουσιάζει ένα υψηλό δυναμικό και είναι μεγάλη η ευθύνη της Ένωσης το δυναμικό αυτό να το χρησιμοποιήσει. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ο Earl of Dartmouth έχει ε, τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. από την... Νομίζω ότι αυτό το οποίο ε, απογοητεύει στην περίπτωση αυτή είναι μια πίεση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπουν όλο και περισσότερες χώρες. Κάποιες πλούσιες χώρες όπως η Ελβετία και η Νορβηγία δεν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουν να τους καπελώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι φτωχές χώρες το θέλουν. 400 ε, εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί μέσω του προϋπολογισμού σε κάποιες χώρες που δεν είναι μέλη της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα παραμένουν σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν προβλήματα και στις χώρες μέλη επίσης. Και από τη δική μου προοπτική έχουμε να κάνουμε με, μια γιγαντιαία αποτυχία αν θέλετε στην προσπάθεια αυτή και ε, πράγματι η Αλβανία στην ουσία θα αδειάσει από τους Αλβανούς που θα πάνε σε μεγαλύτερες και ισχυρότερες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο όπου η κοινωνική προστασία παρέχεται δωρεάν. Ε, τα λέω όλα αυτά ε, και δεν ισχύουν μόνο θα έλεγα στα πλαίσια του αλβανικού θέματος και δεν είναι προς όφελον τελικά της ίδιας της Αλβανίας. Καλό θα είναι η αρμόδια επιτροπή, ο αρμόδιος επίτροπος μάλλον να πει στην Αλβανία ότι δεν πάτε πουθενά έτσι όπως είναι τα πράγματα στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα σας, θέλουμε να είμαστε φίλοι, θέλουμε να σας βοηθήσουμε, αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε και πέραν τούτου ουδέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομο θα είμαι. Εγώ βρίσκω εξαιρετική την πλήρη αυτή η έκθεση του κύριου Κούκαν που νομίζω ότι περιγράφει με σωστό τρόπο το τι θα γίνει τις επόμενες έξι εβδομάδες μέχρι ότου αποφασίσει δηλαδή το Συμβούλιο αν θα χορηγήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας στην Αλβανία. Χρόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πιστούν οι χώρες μέλη ότι μπορούν να ακολουθήσουν τις σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να χορηγήσουν το καθεστώ ε, της ε, υποψήφιας χώρα. Από την άλλη μεριά, το Συμβουλίο δεν έχει λάβει την απόφαση αυτή, ούτε είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η απόφαση αυτή. Κάτι που όμω είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ ακολουθεί νέα διαφορετική προσέγγιση. Ο αγώνας κατά τη διαφθορά, ο αγώνας υπέρ του κράτου δικαίου μπαίνουν ω πρώτε τι προτεραιότητε. Και εν αυτών πρέπει να δει κανεί την ε, διαδικασία ένταξης σαν, μάλλον, την έναρξη διαδικασίας ένταξης σαν μια αρχή μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Μπορεί όμως και να μην ακολουθήσει το Συμβούλιο την ε, σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έκανε για τη Μακεδονία και στην περίπτωση αυτή να δούμε ποιες επιπτώσεις θα έχει ε, στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Κύριε εσείς. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κούκαν ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας θέλει να προσθέσει κάτι επιπλέον. Έχετε το λόγο κύριε Κούκαν. Τίποτα περισσότερο. Καλώς αγαπητοί συνάδελφοι. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το debriefing το οποίο θα μας παρουσιάσει ο συνάδελφος κύριος Λίζεκ για την παρακολούθηση των εκλογών στην Γεωργία στις 27 Οκτωβρίου. Έξι μέλη της Επιτροπής μας υπό την καθοδήγηση του κύριου Λίζεκ στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας συνεργάστηκαν με κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες ε, του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Οι εκλογές γενικά ε, οργανώθηκαν με διαφανή τρόπο, με αποτελεσματικό και επικοδομητικό τρόπο. Ο υποψήφιος που πλειοψήφισε πήρε το 62 περίπου της 100. και είναι κάτι το οποίο εντάσσεται με, με σημαντικό τρόπο στις δημοκρατικές διαδικασίες ε, στην χώρα γιατί υπάρχουν πάντα πολλά τα οποία μέλη να γίνουν. Στην Γεωργία θα πάρει το λόγο ο κύριος Λίζεκ και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στη Γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είχα την χαρά και την τιμή να ηγηθώ της αποστολής παρατήρησης εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Γεωργία. Βέβαια σύντομης, σύντομη ε, επίσκεψη, μόνο τέσσερις ημέρες, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, οι οποίες έγιναν Κυριακή και μία μέρα μετά. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε κυρίως με τους σημαντικότερους υποψηφίους για τις εκλογές. Συναντηθήκαμε και με δημοσιογράφους από διάφορα μέσα ενημέρωσης συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των ε, ε, οργανώσεων των πολιτών της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής με εκπροσώπους άλλων διεθνών οργανώσεων για παράδειγμα με την κοινοβουλευτική, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, επίσης του ΩΣΑ. Η συνεργασία ήταν καλή, δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαστάσεις απόψεων για την αξιολόγηση των εκλογών, εκτός από τις συναντήσεις που είχαμε με τις άλλες αυτές αντιπροσωπείες, ως αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντηθήκαμε την Παρασκευή το βράδυ και με τον αποχωρούντα πρόεδρο Σάκασβίλη και την Κυριακή συναντηθήκαμε, συναντήσαμε με τον νυν πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κύριο Σάμπασβίλη. Χρήσιμες συναντήσεις και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, στον πρώτο γύρο των εκλογών, αυτή έχει, αυτός έχει λήξει τώρα, ο κύριος Αμπασφίλη έλαβε περίπου 62% και λέω περίπου διότι τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται σε λίγες μέρες. Ο δε βασικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης του κόμματος Σακασβίλη δηλαδή, πρόεδρος του Κοινοβουλίου, έλαβε 22%. Το τρίτο αποτέλεσμα ήταν το Μποτανάτζε και ανέρχεται περίπου σε 10% των ψήφων. Υπάρχει και ένας υποψήφιος ακόμη που έλαβε 2 μόλις 100 και ένας άλλος 1%. Όλοι οι υπόλοιποι, 23 ε, συνολικά, έλαβαν στην ουσία μηδενική υποστήριξη. Εδώ επιθυμώ να τονίσω ένα γεγονός. Με τις εκλογές αυτές αλλάζει το πολιτικό σύστημα στην Γεωργία. Από μια Παροεδρευόμενη δημοκρατία τώρα ή μάλλον από μια προεδρική δημοκρατία τώρα μπαίνει περισσότερο σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. 99% των αρμοδιοτήτων του τα εκχωρεί ο πρόεδρος υπέρ του πρωθυπουργού, του αρχηγού της κυβερνήσεως. Πρόκειται για σημαντική μετατόπιση των βαρών στην, της βαρύτητας στο πολιτικό σύστημα. όλες, όλοι οι υποψήφοι και όλα τα πολιτικά κόμματα που συμμετέσχουν θεωρούμε ότι μπόρεσαν να οργανώσουν ελεύθερα τις προεκλογικές τους εκστρατείες, μπόρεσαν να διεξαχθούν πολιτικές συγκεντρώσεις και όπου σημειώθηκαν συμβάντα και υπήρξαν τέτοια, εκεί δηλαδή όπου οι οπαδοί του κυβερνητικού κόμματος προκάλεσαν προβλήματα στους υποψήφιους της αντιπολίτευσης. Ακόμα και ο ίδιος ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης είχε τέτοια προβλήματα. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν αποτελεσματικά και εξασφάλισαν την τάξη και την ασφάλεια. Τα μέσα ενημέρωσης ήταν λίγο πολύ αντικειμενικά, ανεξάρτητα του γεγονότος εάν τα, τα συγκεκριμένα μέσα τάσσονταν υπέρ ενός κόμματος και κατά ενός άλλου. Τα τονίζουμε αυτά βέβαια και στην εκθεσή μας ότι δηλαδή η ενημέρωση ήταν σχετικά αντικειμενική και ιδίω αυτό αφορά τους ιδιωτικούς σταθμούς. Έγιναν και συζητήσεις στις τηλεοράσεις προεκλογικές. Δεν υπήρξαν δηλαδή σημαντικά προβλήματα. Ένα γεγονός το οποίο απασχόλησε και όλους τους διεθνείς οργανισμούς ήταν ένα μειονέκτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και πριν ασκήθηκε ένα είδος πίεσης τους ε, μαχητικούς οπαδούς προκαλώντας προβλήματα σε ορισμένους, σε ορισμένες τοπικές οργανώσεις ορισμένων κομμάτων. Δεν διευκολύνθηκε βέβαια και το ε, πολιτικό κλίμα με την σύλληψη ορισμένων μελών του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού ο οποίος κρατείται. Μπορέσαμε όμως να τον επισκεφθούμε στον τόπο που κρατείται και τον συναντήσαμε τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Φαίνεται η πολιτική κατάσταση μετά τις εκλογές στην Γεωργία να είναι σαφής. Είναι σαφές δηλαδή ότι μπορεί να αναλάβει την κυβερνητική ευθύνη ένα πολιτικό κόμμα που λέγεται το Γεωργιανό Όραμα. Το κόμμα του αποχωρούντος πρόεδρου Σάκασφίλη είναι η δεύτερη σημαντική δύναμη και ο τρίτος υποψήφιος Μποτανάτζε ή μάλλον η υποψήφια Μποτανάτζε ήταν και η μόνη η οποία αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών διότι δήλωσε ότι δεν είχε επαρκή πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, επίσης δεν έλαβε επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή ακούσαμε από την δική της πλευρά κριτικές παρατηρήσεις για την διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας. Στην έκθεσή μας τώρα, επί της οποίας συμφώνησαν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, λέμε, και αυτό ίσως είναι το πλέον σημαντικό, ότι θεωρούμε ότι στις εκλογές αυτές οι Γεωργιανές και οι Γεωργιανοί μπόρεσαν να ψηφίσουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς η, την ίδια την ημέρα των εκλογών δεν σημειώθηκαν δυσκολίες και η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αλλά και οι επιτροπές στις εκλογικές περιφέρειες λειτουργήσαν με υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Ήταν καλά εκπαιδευμένα τα μέλη τους, γνώριζαν τι πρέπει να πράξουν και η όλη διαδικασία ήταν καλά οργανωμένη. Η καταμέτρηση των ψήφων... Ε, κοιτάξτε, εκεί γνωρίζετε ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο, αλλά πάντως ήταν αρκετά αποτελεσματικά οργανωμένοι. Εν τέλει, η αξιολόγησή μας, των διεθνών οργανισμών δηλαδή, είναι θετική. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, señor Lisek. Señor Sigwick. Ευχαριστώ. E, e. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Λίζεκ ε, ξέρει πολύ καλά πλέον ε, το πώς έχει, πώς έχουν τα πράγματα στη Γεωργία και το πολιτικό περιβάλλον, λέει ο κύριος Σίβιακ. Πρόκειται για μια νεαρή δημοκρατία βεβαίως και επομένως ε, καμιά φορά υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Ε, και είδαμε και σε αυτή την περίπτωση στη Γεωργία ότι υπήρξαν κάποιες εντάξεις, εντάσεις, συγγνώμη, ε, οι οποίες εντάθηκαν κατά κάποιο τρόπο και την παρουσία του απερχόμενου Πρόεδρου Σακασβίλη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το εκλογικό σύστημα στην ουσία το επέβαλε ο απερχόμενος πρόεδρος έχοντας την βεβαιότητα τότε ότι θα κέρδιζε τις εκλογές. Αλλά τελικά δεν του βγήκε το πρόγραμμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει έλεγα λοιπόν ότι στη Γεωργία είναι νεαρή δημοκρατία ε, η οποία όμως έχει προοδεύσει ε, αρκετά γιατί βλέπετε ότι εξέλεξαν πρόεδρο με την πρώτη, στον πρώτο γύρο. Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση ε, στις ε, παλαιές σοβιετικές δημοκρατίες ε, να έχουμε τέτοια επιτυχία πούμε, και τέτοια δυνατότητα εκλογής του Προέδρου από τον πρώτο γύρο και με τέτοιο ποσοστό. Τώρα, η συμμετοχή στις εκλογές. Ε, δεν άκουσα στοιχεία από τον κύριο Λίζεκ, αλλά ε, από ό,τι γνωρίζω η αποχή ήταν μάλλον μικρή ε, και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και καλή παρουσία των, και παρουσίαση των υποψηφιωτήτων, καλή δυνατότητα επιλογής από πλευράς των πολιτών με ισότιμες συνθήκες κτλ. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ενισχύεται η δημοκρατία στη Γεωργία, προχωράει προς τη σωστή δημοκρατία και επομένως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο βαθύτερα ίσως το πολιτικό σύστημα που ισχύει στη Γεωργία. Εγώ είμαι ε, εισηγητής για την πολιτική γειτονία και οδηγούμε θα σιγά σιγά και προς μια διάσκεψη ε, κορυφής Ε, και πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές ε, διασταυρώσαμε τα ξύφη μας έχοντας όμως εσφαλμένη άποψη για την πραγματικότητα της γεωργίας. Ε, αναφερόμαστε σε μία σειρά προϋποθέσεων για την χώρα αυτή που τελικά δεν απηχούν την πραγματικότητα. Η γεωργία προσπαθεί πραγματικά να βελτιωθεί, προσπαθεί να προχωρήσει και θα ήθελα τα θετικά αυτά ε, στοιχεία τα οποία ακούσαμε από τον ε, συνάδελφο να ακουστούν και στη της κορυφής του Βίλνιους. Ε, να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για μια θαραλέα χώρα για μια χώρα την οποία θα πρέπει να δούμε με πολύ θετικό μάτι. Όχι μόνο γιατί μόλις ολοκληρώθηκαν εκεί οι εκλογές, αλλά και γιατί η στάση μας ε, ε, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη απέναντι σε μια χώρα η οποία διαρκώς δυναμώνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίβιτς. Η κυρία Νέτς. very much, I would... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον κύριο Λίζεκ για αυτήν την πολύ ενδελεχή ματιά που μας έδωσε για, την, για τις εκλογές στην Γεωργία. Έτσι είχα τη δυνατότητα πριν δύο μήνες να πάω στη Γεωργία και να μιλήσω με τους πρωταγωνιστές και στις εκλογές εκεί. Και εγώ και οι συνάδελφοι μας επισκέφθηκαν επανειλημμένα εκπρόσωποι και του Πρόεδρου Σακασφίλη και πήραμε και τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη χώρα. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από ότι οι εκλογές πήγαν καλά, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται ότι ήταν δίκαιες, ελεύθερες. Μπορούμε βέβαια να ασχολιάσουμε την ηρωνία του ότι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος την οποία πρέσβευε για τον εαυτό του ο κύριος Σάκασβίλη ε, θα γίνει από τον διάδοχό του, ο είναι και ο βασικός του αντίπαλος βέβαια. Αυτό είναι μια ηρωνία της ιστορίας. Πάντως, στα πλαίσια πριν από τη συνάντηση του Βίλνιους, τα πράγματα πήγαν καλά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στη Γεωργία από κοντά γιατί όπως γνωρίζετε ο Πρωθυπουργό δήλωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παραιτηθεί και αυτό φυσικά θέτει ορισμένα σημαντικά ερωτηματικά για το πώς σαν παράδειγμα θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Το ότι πήγαν σκαλά οι συγκεκριμένες εκλογές είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι καθυσυχαστικό αλλά θα ζητήσω από τους συναδέλφους και από το Κοινοβούλιο να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην Γεωργία ε, παρά το ότι πήγαν όπως είπαμε πράγματι πολύ καλά οι συγκεκριμένες εκλογές. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θέλετε εκ νέου το λόγο κύριε Λίζεκ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σύντομα σχόλια θέλω να κάνω. Το πρώτο αφορά τον κύριο Σίβιτς. Δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλη η ε, συμμετοχή στις εκλογές, κάτω από το 50%, αν θυμάμαι καλά 47%. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό, ίσως γιατί οι Γεωργιανοί κατάλαβαν ότι ε, η νέα θέση του Προέδρου θα, είναι, ε, θα έχει λιγότερη βαρύτητα πλέον στο νέο σύστημα και γι' αυτό δεν προσήλθαν στις κάλπες αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε και με τον επικεφαλής, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ότι δηλαδή υπάρχει και μια ένα σχετικός εκνευρισμός ε, στην ε, κυβέρνηση ε, για την, διαφο... για την έτσι, τροποποίηση του συστήματος. Ε, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος, ο περχόμενος πρόεδρος Σακασβίλη έχει χάσει τις εκλογές ε, και ο πρωθυπουργός Ιβανισβίλη θα ε, παρετηθεί. Στην ουσία θα παρατηθεί στο τέλος αυτού του μήνα. Έχει οριστεί ένας νέος πρωθυπουργός, ο οποίος ενδεχομένως ε, θα ε, ε, υπερψηφιστεί, δηλαδή θα έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, αλλά που δεν θα είναι το ίδιο δυνατός με τον προηγούμενο, γιατί είναι ένας πολύ νέος πολιτικός, 31 ετών, νέος και στην πολιτική σκηνή της Γεωργίας. Από την άλλη πλευρά βέβαια ίσως είναι καλό που είναι νεαρός. Παραμένει πάντως γεγονός ότι δεν θα έχει τόσο πολύ δυνατή θέση στην κυβέρνηση είναι νέος πολιτικός και ο πρόεδρος ε, προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο, είναι φιλόσοφος, αυτό είναι το επαγγελμά του. Και επομένω θα έχουμε νέο πρόεδρο και νέο πρωθυπουργό ε, και οι δύο όμως είναι άγνωστες πολιτικές ε, προσωπικότητες. Παραμένουν λοιπόν όντως κάποια ερωτηματικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ με την παρέμβαση αυτή. Κλείνουμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. Θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο το οποίο έχουμε να συζητήσουμε για σήμερα, το debriefing που θα έπρεπε να κάνει η Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας της Αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης μετά την συνάντησή στις 20 Οκτωβρίου στη Γάζα. Δεν είναι εδώ η πρόεδρος, αλλά ο κύριος Σάτκινς ε, μας περιμένει με υπομονή και του δίνουμε τώρα τη δυνατότητα να μας ενημερώσει. Κοιτάξτε, είπα ότι θα μπορούσα να σχολιάσω ε, την αντιπροσωπεία αυτά ε, λόγω της απουσίας γενικά και του Προέδρου μας επειδή έχει μειωθεί και η ημερήσια διάταξη ίσως να ήταν χρήσιμη η παρουσίασή μου. Αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ενέργεια εναντίον της κυρίας Κοστέλο, η οποία θα κάνει την παρουσίαση που πρέπει όταν πρέπει. Πάντως νομίζω ότι το θέμα θα ενδιαφέρει τους συναδέλφους. Είμαστε η επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στη συνάντηση ε, με το Συμβούλιο το Παλαιστινιακό έπρεπε να συναντηθούμε στη Γάζα. Δεν μπορέσαμε να πάμε στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια. Ψηφίσαμε βέβαια 300 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια και ήμασταν πάρα πολύ θυμωμένοι γιατί οι Ισραηλινές αρχές μας απαγόρευσαν για μια ακόμη φορά από το να πάμε στη Γάζα μέσω από το πέρασμα του Χερέτς το οποίο είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να πάμε λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο πέρασμα Ραφά στην, στην νότια πλευρά της Γάζας, στα σύνορα με, της Αίγυπτο, την Αίγυπτο. Ε, υπάρχουν θέματα και στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στο Μεσανατολικό. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο εμένει στις θέσεις αυτές και το Ισραήλ επέμενε και αυτό με τη σειρά του και δεν μας άφησε να πάμε και γι' αυτό φτιάξαμε ένα πρόγραμμα ε, για τη δυτική όχθη μόνο ε, είχαμε την καλή τύχη να συναντηθούμε με τον νέο Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, παρά τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και επίσης τον Υπουργό για τις φυλακές, ο οποίος μας είπε το τι συμβαίνει στην ε, περίπτωση του δικού του τομέα. Και υπήρξε απελευθέρωση 27 ε, κρατουμένων, πάρα πολύ δημοσιότητα δόθηκε σε αυτό θα ήθελα να πω ότι αν δεν είναι κανείς πάρα πολύ κοινικός, ναι μεν 26 απελευθερώθηκαν, παραμένουν όμως, ε, ε, ανακοινώθηκαν όμως 1.700 νέες προσπάθειες επικισμού και ταυτόχρονα μέσα σε 24 ώρες υπήρξαν άλλοι 26 οι οποίοι συνελήφθησαν από τις δυνάμεις κατοχής. Συνεπώς η απελευθέρωση των συγκεκριμένων προσώπων δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό και από τον ανώτερο διαπραγματευτή της Παλαιστινιακής Αρχής ε, τι πρόοδος έχει υπάρξει σε σχέση με τις δραστηριότητες ε, του ε, Υπουργού Εξωτερικών κ. Κέρι. Τα πράγματα μας είπαν πάνε καλά. Όταν τους είπαμε πιστεύετε πράγματι ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή, η βασική απάντηση ήταν μπα. Αυτό έγινε γιατί το Ισραήλ συνεχίζει να χτίζει νέες, ε, ε, νέες εγκαταστάσεις, νέους οικισμούς και οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι από τις συνθήκες αυτές. Ήρθαμε σε επαφή και με τους εκπροσώπους της Σόκρα των Ηνωμένων Εθνών να πω ότι οι εκπρόσωποι των ΗΕ υψηλοπάτου επίπεδου είναι πάρα πολύ αντικειμενικοί, βαθείς γνώστες της κατάστασης και μας καθοδήγησαν και σε σχέση με τις δραστηριότητες της Ούνρα και σε σχέση με τις δραστηριότητες της Όκρα και για τις εγκαταστάσεις δηλαδή και για την προσπάθεια βοήθεια σε τρόφιμα κτλ. Ε, η πρώτη γραμμή της Ισραηλινής πολιτικής είναι 5.000 νέοι οικισμοί που θα ξεπεράσουν τη Βόρεια Ιερουσαλήμ και θα διαιρέσουν τη δυτική όχθη σε δύο τμήματα ε, στην ουσία καθιστώντας αδύνατη τη λύση των δύο, ε, ενός κράτους δύο κρατών ε, πραγματοποιήσιμη. Υπάρχουν και τα προβλήματα με τους Βεδουίνους, μας είπανε το από πού εξεδιώχθησαν οι Βεδουίνοι έτσι ώστε να ξεκινήσουν αυτές ε, οι οικοδομές. Ανησυχούμε λοιπόν για την απομάκρυνση τη βία των Βεδουίνων και για τους οικισμούς των Ισραηλινών. Μας είπαν ότι υπάρχει επίσης και σκόπιμη πρόκληση βίας από πλευράς των επίκων και εκεί που συναντηθήκαμε με τους Βεδουίνους, οι οποίοι νόμιμα ήταν στον τρίτο τομέα, ένας από τις δυνάμεις ασφαλείας με κάμερα και ε, γενικά όπλα πολλά ήρθε και μας απείλησε επειδή υποστηρίζουμε αυτούς οι οποίοι απομακρύνονται δια της βίας από τους χώρους κατοικίας τους. Ξέρω πρόεδρε ότι θέλετε να προχωρήσετε τη συζήτηση, να πω ότι τα δύο πράγματα τα οποία βασικά μάθαμε και ξέρω ότι η πρόεδρός μας ε, είναι σε επαφή και με τους κοσμήτωρες σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στη Γάζα και τα εμπόδια της Ισραηλινής κυβέρνησης. Να πω ότι συναντηθήκαμε εμείς και με τον κύριο Τζον Γκατράτα, τον οποίο είχαμε συναντήσει και εδώ και ο οποίος αυτός είναι επίσης υψηλής ποιότητας εκπρόσωπος και εκτιμάται δεόντως από τις τοπικές αρχές. Ε, και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους εκπροσώπους του κουαρτέτου, ε, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει με το κουαρτέτο στα πλαίσια των καθημερινών τους ε, επαφών με τα ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές δεν έχουν καθόλου μα καθόλου καλές σχέσεις, δεν τους εκτιμούν καθόλου. Είχαμε όμως τις ανησυχίες του Υπουργού των Φυλακών που μας είπε ότι οι Ισραηλινοί δοκιμάζουν, κάνουν ε, ε, τεστ, πειράματα με φάρμακα στους Παλαιστινίους, στις, Παλαιστινιακές, στις Ισραηλινές φυλακές. Αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο, δεν σημαίνει τίποτα η λέξη απαράδεκτο, είναι πραγματικά εκρηκτικά απαράδεκτο. Όπως φαντάζεται κανείς οι Ισραηλινοί δεν σέβονται τη σύμβαση της Γενέβης ή τα διεθνή δικαιώματα, αλλά σύμφωνα με τον στρατιωτικό τοπικό νόμο. Συνεπώς κάνουν ό,τι τους καπνίσει γενικότερα. Οι συνάδελφοι λοιπόν κατανοούν ότι υπάρχει επίσης ένα αίτημα από υψηλό αριθμό μελών να επισκεφθούν και να ελέγξουν τις φυλακές και τους φυλακισμένους. Ο Υπουργός λέει είναι πέντε αστέρων οι φυλακές μας οι καλύτερες φυλακές στον κόσμο και ταυτόχρονα όμως μας εμποδίζουν να πάμε να τις επισκεφθούμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής μας να ελέγξουμε τις φυλακές αυτές και αυτό είναι μία επιπλέον αντίφαση για την οποία θα πρέπει να ανησυχούμε. Και τέλος κύριε πρόεδρε, συνειδητοποιούν οι συνάδελφοι ότι υπάρχουν 200 περίπου παιδιά κάτω των 17 ετών στις Ισραηλινές φυλακές. Όταν πηγαίνουν επισκέπτες στις φυλακές αυτές ε, τους παρουσιάζουν όλους ανά 30 σε τάξεις. Κατά τα άλλα είναι μοιρασμένοι με τους ενήλικες και κανένας δεν ασχολείται ειδικά μαζί τους. Και το ίδιο ισχύει επίσης και για τους 100 φυλακισμένους εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι οποίοι πεθαίνουν από τερματικές μορφές ε, ε, καρκίνου και οι οποίοι το μόνο που τους δίνουν είναι παρακεταμόλοι. Ε, για να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος στις φυλακές των Ισραηλινών. Λοιπόν, ε, όλα αυτά ξέρω ότι η Πρόεδρος θα σας τα πει λεπτομερέστερα και ο Πρωθυπουργό και όλοι μας είπαν όπως πολύ συχνά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία το μόνο που κάνει είναι να δίνει λεφτά, να καλύπτει τα έξοδα ε, αυτό το κάνει για να καθησυχάσει τις συνειδήσεις, αλλά δεν παίζει κάποιο ρόλο έτσι ώστε να υπάρξουν εκλογές, να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, να τεθεί τέλος στη βία, στους οικισμούς κτλ. Γιατί δεν παίζουμε έναν μεγαλύτερο ρόλο. Δεν το κάνουμε λοιπόν αυτό και οι Παλαιστίνοι τους οποίους συναντήσαμε, οι οποίοι μόνο τρομοκράτες δεν είναι, εξέφρασαν την μεγάλη τους λύπη για την έλλειψη του ρόλου αυτού και την ελπίδα ότι κάποτε θα το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά περίπου ε, νιώσαμε και αισθανθήκαμε εκεί στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα ενημέρωση κύριε Άτκινς. Όπως είπατε πολύ σωστά θα συνεχιστεί η παρουσίαση αυτή δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση τώρα γύρω από τα θέματα αυτά, τη απουσία της Προέδρου της Επιτροπής, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σίβιτς, αλλά σύντομα παρακαλώ. Αυτή η συζήτηση δεν θα αντικαταστήσει την συζήτηση ε, που θα ακολουθήσει. Κάνουμε τη συζήτηση αυτή επειδή το ζήτησε ο κ. Σάτκινς. Το θέμα είναι μεγάλο, το θέμα είναι σημαντικό και θα γίνει συζήτηση στο επίπεδο το οποίο προβλέπεται την παρουσία της Προέδρου της Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κ. Σιβίτσου. Ναι, βεβαίως. Δεν έχω καθόλου την πρόθεση να ξεκινήσω συζήτηση, άλλωστε είμαστε πολύ λίγοι στην αίθουσα. Μια ερώτηση μονάχα για τον Σερ Ρόμπερτ Άτκινς. Σε ποιο πλαίσιο ε, θέλησε να επισκεφθεί την Γάζα η αντιπροσωπεία, ε, μια ε, ζώνη η οποία δεν είναι η αυτόνομη Παλαιστινιακή ζώνη, αλλά έχει ε, ηγείται πλέον της περιοχής αυτής μια επαναστατική κυβέρνηση η οποία πήρε τη θέση μιας νόμιμη εκλεγμένης κυβέρνησης, ο κ. Ράτκινς. Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να πάμε στην Γάζα είναι γιατί η ε, ε, γιατί εμείς πήγαμε επιλεγμένοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έτσι ώστε να ε, κάνουμε έναν ανθρωπιστικό έλεγχο, να δούμε με ποιο τρόπο σπαταλιώνται, διεξοδεύονται τα χρήματά μας στην Γάζα. Είχαμε αντιπροσωπεία ε, από πολλές πολιτικές ομάδες. Θελήσαμε να έρθουμε σε επαφή με εκπροσώπους πολλών πολιτικών ομάδων έτσι ώστε, ε, άλλωστε και αυτός είναι ο στόχος μας, να δούμε, να ελέγξουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ευχαριστούμε πολύ, ε, Σεράτκιν. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή, η οποία θα συνεχιστεί την παρουσία της αρμοδίας Προέδρου της Αντιπροσωπείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλα θέματα και επομένως λίγη συνεδρία. Ευχαριστώ.